if you take seats and the Καθίστε παρακαλώ. The report is a for Πρώτη έκθεση είναι πρόταση οδηγίε για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτικά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής η λεγόμενη πρόταση της Ευρωβινιέτας. Ξεκινούμε με την τροπολογία 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 108. Έγκρινεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ξεκινούμε την τροπολογία 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. μαζί με τον 125 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ότι 17 άρχεται πέρας απορρίπτεται Πάμε στη 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα σε ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Λέει πρόεδρος. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 και 145 και 146 και 147 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Α, τυχερή ήμουνα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 Περ. κατά, αποχές, ξανά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 Περ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161, 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, μαζί με τα 167 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ...168 και 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 172-173 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 195 με την 181 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε όμως. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 και 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν επόμενε. 35 έως 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπήρξε σύγχυση για την προηγούμενη τροπολογία. Να ξανακάνουμε την 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 πέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 και 205 πέρ κατά. Το ΕΛΚ τι λέει για τις 42 και 205 πέρ κατά. Δεν θέλετε να μου δείξετε.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 211, 13, 14, 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Α, και 212 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 217 και 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 44 και 218 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές απο... απορρίπτεται. Δεν ε, είδα. 226 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 29, 30, 31, 32, 33 και 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 1 άρχεται πέρας εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 55. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 56. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Ναι γιατί υιοθετήσαμε μια συμβαστική πριν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 και 70 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε την 8. Πέρας. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 76. Πέρας. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία κιόλα, αλλά δεν το είχα καταλάβει πριν. Εβδομήντα υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 85, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 86, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 87, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 88, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 89, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές Εσείς είστε κατά. Ξανά. Για την 95. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Next one. Πάμε στο επόμενο. Ψηφίζουμε την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016. Έκθεση πρωτοβουλία συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 7 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 8 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, 9, ας τσεκάρουμε την 8, ηλεκτρονικά. Αποσύρετε το αίτημα, υιοθετείται. Γιατί και το ΕΛ και, το... και οι σοσιαλιστές υπερψήφισαν. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 12 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τη 12. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 3 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. 1 Κατά. Αποχές Ελέγχουμε την 30. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά εποχές Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Και τώρα ψηφίζουμε την ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του προγράμματος LIFE. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθε... Α, Τη 15 δεν την ψηφίζουμε. Δεν την ψηφίζουμε. Χωριστή ψηφοφορία στη 16. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 28 λέει η ε, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 30 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 29 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται, 32 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται, 33 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 34 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε κρονικά 34. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, 39 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 40 υπέρ κατά, α, καταπίπτει, 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 43 υπέρ Σαράντα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ, κατά, αποχές διοθετείται. 46 δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε χρονικά το δεύτερο τμήμα της 46. Πέρας οφορίας. Απορρίπτεται. 47 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν είμαι σίγουρη. Υιοθετείτε. 48. Η πρόταση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 54 ηλεκτρονικά. Είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Όχι λάθος. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοφορίας υιοθετείται 61 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 68 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 69 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 70 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 71 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 3 υπέρ κατά υπέρ της 3 κατά ελέγχουμε ερχονικά την 3 Πέρας. Υιοθετείτε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 όχι. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Ολοκληρώσαμε εδώ τις ψηφοφορίες και τώρα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Σέικχαουτ. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για το πρασίνισμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. απορροφή. Okay, uh, dear colleagues, if you can... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τη σημερινή μας εργασία. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τον προγραμματισμό αυτός και την ειδική έκθεση για το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Είναι τμήμα της ε, ετήσιας ε, δραστηριότητας ε, ελέγχου και των τακτικών σχέσεων που έχουμε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τους προσκαλούμε λοιπόν σε μια κοινή συζήτηση. Έχουμε τα μέλη τους, του ΕΚΑΣ που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις δύο ειδικέ εκθέσεις. Έχουμε τον υπεύθυνο για το πρασίνισμα της ΚΑΠ εδώ και τον κύριο Γιάννους Χοϊφσκόφσκι που είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα τη υπαίθρου, την ανάπτυξη, της ανάπτυξης υπαίθρου. Κύριε Γιάπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία για να παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα και τις, τα συμπεράσματα από την ειδική έκθεση «Το Πρασίνισμα», ένα πιο περίπλοκο σύστημα στήριξης του εισοδήματος που δεν είναι ακόμα ε, περιβαλλοντικά αποτελεσματικό. Το πρασίνισμα εισήχθη το 2013 με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ως ένας ε, μηχανισμός άμεσων πληρωμών στους ε, γεωργούς. Ε, σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός για να ανταμείψει τους γεωργούς για τα δημόσια αγαθά που προσφέρουν και να ενισχύσουμε τις ε, περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΑΠ. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το πρασίνισμα που είναι 30% όλων των άμεσων πληρωμών της ΚΑΠ και το 8% ολοκλήρου του προπολογισμού. οι γεωργοί λαμβάνουν την έλαβαν την πρώτη τους πληρωμή για το πρασίνισμα το 2016 για τις αιτήσει του 2015 γενικά, όμως, οι προϋποθέσεις αυτές, ε, τα βασικά μας προβλήματα μάλλον από, το, την έκθεση, είναι ότι είναι απίθανο να έχουμε ουσιαστικές ε, βελτιώσεις στις επιδόσεις περιβαλλοντικές και κλιματικές της ΚΑΠ. Οι προποθέσει του πρασινίσματο γενικά ε, ε, είναι προβληματικές, ε, δεν δίνουν αποτελέσματα και γενικά ε, δεν απεικονίζουν, τις, απεικονίζουν απλώς τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές. Έχουμε ουσιαστικές εξαιρέσεις, περισσότεροι γεωργοί, το 65% αποφελούνται από την πράσινη πληρωμή, χωρίς ουσιαστικά να υπόκεινται σε ειδικέ υποχρεώσει του πρασινίσματο. Ω αποτέλεσμα, το πρασίνισμα ε, οδηγεί σε θετική αλλαγή στι ε, γεωργικέ πρακτικέ σε πολύ περιορισμένο αριθμό των περιπτώσεων, ένα 5%. Εμείς χρησιμοποιούμε ε, ένα βασικό δείκτη, το το 73% της γεωργικής γης ε, έχει τουλάχιστον μία υποχρέωση πρασινίσματος. Ακόμα και αν η εκμετάλλευση υποχρεούται να ακολουθήσει τις προϋποθέσεις για την διαφοροποίηση των καλλιεργειών και να αλλάξει τις καλλιέργειες, στην πραγματικότητα αλλάζει μόνο το 1 εκτάριο από τα 100 εκτάρια και η Κομισιόν παρόλα αυτά μετράει και τα 100 εκτάρια με βάση αυτό το νούμερο όλο το μέγεθος εκμετάλλευσης ε, συνυπολογίζεται υπό αυτό το δείκτη και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στι γεωργικές πρακτικέ, γιατί ο γεωργός ουσιαστικά σέβεται, σεβό, ε, σεβόταν ε, τους κανόνες του πρασινίσματο πριν εισαχθεί το πρασίνισμα. Αυτό ο δείκτης δεν θα αλλάξει. Ακόμα και αν υποχρεώσει υπό το πρασίνισμα ε, αλλάξουν ουσιαστικά. Παραδείγματο χάρη η ΕΦΑ που αν καλύψουν 3 ή 5 ή 7% δεν αλλάζει τίποτα. Βρήκαμε λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν έχει θέση συγκεκριμένους στόχους ή δεν έχει προσδιορίσει τι αναμένουμε να πετύχουμε μέσω του πρασινίσματος ε, για το περιβάλλον και το κλίμα. Η περιβαλλοντική και κλιματική επίπτωση του πρασινίσματος συνδέεται με την ε, θεματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του εδάφους που αφορά την ποιότητα του εδάφους. το παρκέτο Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 για το κλίμα και την ενέργεια και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια του 2030 ε, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα και την στρατηγική βιοπικιλότητα. Χωρίς να θέσουμε όμως συγκεκριμένους στόχους για την ΚΑΠ, δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική προσέγγιση για να υλοποιηθούν αυτές τι στρατηγικές. Οι συζητήσεις για το πρασίνισμα δεν θα πρέπει να κινούνται γύρω από το ερώτημα του αν το πρασίνισμα ουσιαστικά ήθελε να ενισχύσει τις επιδόσεις περιβαλλοντικές ή να μειώσει την ε, υποβάθμιση των περιβαλλοντικών δικτών. Κοιτάξτε, ας πούμε, έναν δίκτυο. ας πούμε. Ε, ο δίκτυς για τα πτηνά στις α, ε, γεωργικές γεές μειώθηκε κατά 31,5% από το 90% στο 2014. Το βασικό ερώτημα δεν είναι ε, κατά πόσον πρέπει να βελ... δεν είναι το κατά πόσον πρέπει να βελτιώσουμε τους, α, τις περιβαλλοντικές περιπτώσεις της, της ΚΑΠ. Είναι πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχουμε βασικά στοιχεία. Η κατανομή του προπολογισμού για το πρασίνισμα δεν δικαιολογείται από το περιεχόμενο τη περιβαλλοντική πολιτική. Ε, οι πληρωμέ του πρασινίσματο είναι 80 ευρώ το αναεκτάριο ε, και στη μελέτη αντικτύπου εκτιμάται ότι το μέσο κόστο για την εφαρμογή των μέτρων πρασινίσματο ε, δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 30 ευρώ. Στην πραγματικότητα το πρασίνισμα και οι πληρωμέ αυτέ είναι για να στηρίξουν τις πρέπει να στηρίξουν ουσιαστικά τις γεωργικές πρακτικές. Ε, το, του πρασινίσματος ουσιαστικά είναι ένα σύστημα στήριξης του εισοδήματος. Οι περιορισμοί στο σχεδιασμό μειώνουν την αποτελεσματικότητα τριών πρακτικών. Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν ε, δίνει πλήρη περιβαλλοντικά ωφέλη και δεν δίνει τόσο ωφέλη όσο θα δίνει η άμυψη σπορά. το ESPG ε, δηλαδή, οι μόνιμα ευαίσθητες, ε, τα μόνιμα ευαίσθητα βοσκοτόπια έχουν σχεδιαστεί άσχημα και δεν στοχεύουν τις, ε, τους βοσκότοπους που έχουν πολύ μεγάλο απόθεμα σε άνθρακα, εκτός του Natura 2000. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν την ευελιξία για την εφαρμογή του πρασινίσματος, ειδικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των ειδών ΕΦΑ και τον καθορισμό των περιβαλλοντικά ευαίσθητων μόνιμων βοσκοτόπων για να βελτιώσουν, για να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη της πολιτικής στο κλίμα και το περιβάλλον. Εφαρμόζουν απλώς ε, το πρασίνισμα για να μειώσουν όσο μπορούν το βάρος στο, στα ίδια και στους γεωργούς. Με βάση αυτά τα πορίσματα κάνουμε τις, επόμε... τις ακόλουθες συστάσεις για την επόμενη ΚΑΠ. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναπτύξει μία πλήρη λογική παρέμβαση για τη συνεισφορά της ΚΑΠ στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακολουθούν αυτές οι, οι αρχές, δηλαδή και ποιες είναι αυτές, ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γεωργοί στις πληρωμές ΚΑΠ μόνο εάν πληρώνουν ε, μια βασική δέσμη περιβαλλοντικών κανόνων που καλύπτονται από τις τρέχουσες πρακτικές βέλτιστε γεωργικές πρακτικές της ε, ΓΑΕΚ και το πρασίνισμα. Και επίσης, ειδικέ ε, και, περιβαλ... και τοπικές περιβαλλοντικές και κλιματικέ ανάγκες ε, αντιμετωπίζονται μέσω από ισχυρότερα προγράμματα και δράσεις και ανταμείβονται οι γεωργοί για υπηρεσίε που ξεπερνούν τι βασικέ περιβαλλοντικέ υπηρεσίε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποδεικνύουν πριν από την εφαρμογή ότι οι συγκεκριμένε επιλογέ που διαλέγουν είναι αποτελεσματικέ. Επίσης, θα ήθελα ε, να πιστεύω ότι ε, με την τελευταία νομοθεσία Omnibus θα έχουμε κάποιες βελτιώσεις, γι' αυτό είναι, είμαστε θετικοί απέναντι σε αυτή. Αλλά υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την απλούστευση και τις καλύτερες ε, επιδόσεις του πρασινίσματος που πρέπει να επιληθούν στο επόμενο πολιτεύσιμο πολιτισμό-συνομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αν έχετε ερωτήσεις να σας απαντήσω. Θα κάνετε και εσείς την παρουσίασή σας. Thank you very much, uh, Madam President, uh, uh, distinguished members of... Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ε, πρόσκλησή σας και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση με τίτλο ε, «Προγραμματισμός της ανάπτυξης της υπαίθρου επικεντρωνόμενη στα αποτελέσματα». Όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και από άλλε εκθέσει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε συνεργεί για την ανάπτυξη υπαίθρου και την περιβαλλοντική πολιτική και άλλε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και σα ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον προγραμματισμό της πολιτικής ανάπτυξη υπαίθρου. Όπω και ο θα χρησιμοποιήσω και εγώ τι διαφάνειε για να σα κάνω την παρουσίαση. Ε, τι είναι, σημαίνει με τον προγραμματισμό της πολιτικής ανάπτυξη υπαίθρου. Βλέπετε τις δαπάνες ε, για τον προγραμματισμό ε, για την επταετή περίοδο 100 δις. Βλέπουμε πως υπάρχουν τα διάφορα τμήματα της αγγελικής πολιτικής 58 δις ε, το χρόνο, 40 είναι ε, για τις άμεσες πληρωμές, 14 ε, για τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου και 4 για τις, τα όργανα που χρησιμοποιούμε για την αγορά. Επόμενη διαφάνεια. Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι, ποια κράτη-μέλη και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν ε, στο, τομέο, στο ταμείο αυτό η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία όπως βλέπετε είναι, έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Σε αυτό το χάρτη βλέπετε τα προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου ανακράτος μέλος που έχουμε διεξάγει ήδη τους ελέγχους γιατί ο προγραμματισμός για την πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου σε κάποια κράτη-μέλη οργανώνεται σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, έχουμε 118 RDPs ε, σε 28 κράτη-μέλη, ε, περιφέρειες προφανώς εννοεί ο μιλητής, και έχουμε ελέγξει τις 12 από αυτές. Ε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δύο προγράμματα έχουν συμβάλει σε καλύτερα αποτελέσματα, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα και ακριβώς πώς ήταν η περίοδος προγραμματισμού και η διαδικασία προγραμματισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εξετάσαμε. Και ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα. Παρά ήταν γενικά τα προγράμματα, η διάρκεια τους και η περιπλοκότητά τους ήταν ε, υπερβολικές. Ε. Και επίσης δεν υπήρχε κατάλληλη εστίαση. Τι σημαίνει ε, ότι ήταν πολύ γενικά. Δύο παραδείγματα. από τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ιρλανδία. Τρία παραδείγματα. Υπήρχε ασάφεια στον προσδιορισμό των αναγκών. Επόμενο συμπέρασμα ε, ήταν υπερβολικά περίπλοκα τα έγγραφα και η διάρκεια ήταν υπερβολική. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, ε, στην προηγούμενη περίοδο οικονομικών προοπτικών, μέχρι το 2013 δηλαδή, ε, το μέσο μέγεθος ο μέσο όγκος εγγράφων μάλλον του, του προγράμματος ήταν 459 σελίδες, στην επόμενη 781. Και σε, κάποια, σε περίπτωση κάποιων προγραμμάτων πάνω από χίλιες. Όχι pictures στο διάσταση Σελίδε σελίδες εννοούσα. Άνω, άνω λοιπόν των χιλίων σελίδων. Κάποια προγράμματα. Συμπέρασμα. Περιμένει πολλά, υπερβολικά πολλά, Επιτροπή από τις περιφέρειες και από τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά δεδομένα, πολύ χρήσιμα για τις επιστημονικές συζητήσεις, αλλά όχι για τους γεωργούς γιατί είναι υπερβολικά περίπλοκα. Δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό προτείνουμε να αλλάξει αυτό. Να μην υπάρχουν τόσο πολλές απαιτήσει. Και επίσης η εξαιρετικά παρατεταμένη προγραμματική ε, περίοδος προγραμματισμού. Πάνω από 11 μήνες, ένας χρόνος, κατά μέσο όρο. από την ε, αρχική υποβολή μέχρι τις, ε, την επιστολή προς, με τις παρατηρήσεις μέχρι την τελική υποβολή προς την Επιτροπή. ποια, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια ότι άργησε πολύ η εφαρμογή. Σε σχέση με το 2007-2013, η πρώτη πρόταση ήταν το 2004, τα μέτρησα του 2004 επευλήθηκε η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φτάσαμε μέχρι τα τέλη του 2006. Μετά υπήρχε περαιτέρω καθυστέρηση. Τον Οκτώβριο του 2011 για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2014-2020. Και φτάσαμε τον Ιούλιο 2014 μαζί με τον εφαρμοστικό κανονισμό. Επόμενη διαφάνεια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στην περίοδο 14-20 τα τέλη του 2010 μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής, μάλλον είναι στην περίοδο 2007 με 13 ομιλητής, το ποσοστό απορρόφησης ήταν 29%. Στην τρέχουσα ε, περίοδο 2014-20. Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογή, στα τέλη του 2017 δηλαδή, η απορρόφηση ανήλθε μόνο στο 21%. Επόμενη διαφάνεια. Επίπεδο απορρόφηση ε, για την περίοδο 2007-2013. Ο μέσο όρο ήταν 29% όπως σας είπα. Δύο κράτη-μέλη με ε, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο πάνω από 50% ήταν η πρώτη. Και κανείς δεν έπεσε κάτω από το 15% τώρα, στην τωρινή, στην τρέχουσα περίοδο. Είναι, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Ε, μέσος είναι το 21% απορρόφηση. Πρώτη είναι η Φινλανδία, 43%, η Ιρλανδία 38%. Κανείς δεν έχει πάνω από 50% και έχουμε 6 κράτη-μέλη ε, με απορρόφηση κάτω από το 15%. Ε, θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Το επόμενο συμπέρασμα ελέγχου. Ποια είναι η συμβολή των μονομένων προγραμμάτων στρατηγικούς, στην επίδευση στρατηγικών στόχων της Ευρώπης 2020. Δύσκολο να αποτιμηθεί αυτό ποιοι θεματικοί στόχοι έχουν ε, σημασία και ειδικό βάρο για την περιβαλλοντική διάσταση τη ανάπτυξη υπαίθρου, ώστε να υποστηρίξουμε τη μετάβαση προ την ε, οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα σε όλου του τομεί, ε, προσαρμογή για το κλίμα, πρόληψη κινδύνου, διαχείριση, προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεσματικότητα των πόρων. Τι προτείνουμε εμείς προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει μεγαλύτερη σύμφωση μεταξύ των θεματικών προγραμμάτων και άλλων στρατηγικών προγραμμάτων ε, να συνεχίσει να παρακολουθεί και να μετρά τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ε, τους κατάλληλους δείκτες να απλουστεύσει το περιεχόμενο και να μειώσει κυρίως τον αριθμό των απαιτήσεών της. Προτείνουμε επίση να προετοιμάζει τις νομοθετικές προτάσεις για την πολιτική ανάπτυξη του για την περίοδο μετά το 20 εγκαίρως. για να ε, καταστεί δυνατή η έγκριση στην αρχή της προγραμματικής περίοδου. Πρόεδρε, αλλά δύο λεπτά. Επιτρέψτε μου. Στις γενικέ ε, παρατηρήσει για το πρόβλημα, για το γεωργικό τομέα. Γιατί πιστεύω ότι αυτά που θα σας πω είναι πολύ σημαντικά Ε, για το περιβάλλον. Υπάρχουν πληροφορίες ότι βάσει συγκεκριμένων δεδομένων την τελευταία δεκαετία για το εμβαδό της γης που δηλώθηκε ε, μειώθηκε από τα 164 εκατομμύρια εκτάρια, ε, κατά 19 εκατομμύρια εκτάρια μειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Έπεσε στα 145 και ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσα σε 7 χρόνια 3 εκατομμύρια. Την τελευταία δεκαετία χίλιες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις την ημέρα χάνουμε. Αυτός είναι ο ρυθμός ε, μείωσης ε, των ε, μικρών αγροκτημάτων. Η γύρανση του πληθυσμού των γεωργών. Αυτό το γράφημα βλέπετε ότι η μέση συμμετοχή της νέας γενιάς όπως χαρακτηρίζεται, δηλαδή κάτω των 45, 40%, κάτω του 40% ενώ στην οικονομία γενικότερα, στην οικονομία γενικότερα είναι 50% ενώ στη γεωργία είναι μόνο 20%. Ε, ε, ένα τρίτο των γεωργών, όχι, ένα τρίτο γεωργών είναι πάνω από 65 και η μισή γεωργή είναι πάνω, άνω των 45 ετών. Μεγάλο πρόβλημα σας Λοιπόν, βλέπετε την ε, κατανομή, γιατί έχουμε και την έκθεση για τους νέους γεωργούς, ε, την εκπονήσαμε το 2017. Βλέπετε την κατανομή ένα κράτος μέλος. Άλλο ένα μόνο στοιχείο που νομίζω θα είναι σημαντικό για σας είναι ε, νέο έγγραφό μας παρουσιάζουμε αυτά τα δεδομένα και ε, το, την περασμένη εβδομάδα το παρουσιάσαμε στην Επιτροπή ε, Ελέγχου των Προεπολισμών από τον συνάδελφο Ζωά Φιγκρέντ. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι η γεωργική παραγωγή είναι σε καλή κατάσταση γιατί είμαστε καθαρός εξαγωγέας, έτσι, γεωργικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εξάγουμε περισσότερα τρόφιμα από ό,τι εισάγουμε. Μπράβο. Για δείτε, το πράσινο κομμάτι είναι αγαθά και άλλα πρωτογενή προϊόντα. Μη μεταποιημένα δηλαδή εννοώ. Ε, μη μεταποιημένα τρόφιμα. Όμω όμως δεν είναι ε, success story αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι η γεωργική παραγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές μεταποιημένων, όχι στη δική μα παραγωγή. Πρέπει να το λάβετε υπόψη τώρα που προετοιμάζετε τη μελλοντική ε, γεωργική πολιτική. Τελειώνω, Πρόεδρε. Το πρόβλημα ε, που εντοπίζουμε σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο που θα σας παρουσιάσουμε και στο μέλλον είναι ότι χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη ε, θεώρηση, ε, ένα, ένα όραμα για την ε, κοινή γεωργική πολιτική πέραν των 7 ετών της προγραμματικής περίοδου. Μόνο έτσι θα εκπονήσουμε μια καλή γεωργική πολιτική. Χρειάζεται όραμα μακροπρόθεσμο. Πόση οι γεωργοί, πιο ευαδόγοι σε ποιες εκμεταλλεύσεις, μικρές, μεγάλες, τι είδους γεωργία. Μακροπρόθεσμους στόχους χρειαζόμαστε, προτού τοποθετηθούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Thank you very much. Thank you both for your presentation. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Το λόγο έχουν τώρα οι συνάδελφοι. Η κυρία Γιούσο πρώτη. Γερμπράντη, Σαρπέκ. Παρακαλώ, κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Το ελεγκτικό συνέδριο κάνει μία ανάλυση με νούμερα όπως πρέπει να κάνει ένα ελεγκτικό συνέδριο. Και επικρίνει το γεγονός ότι το 71% των γεωργών δεν λαμβάνουν υπόψη το πρασίνισμα. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε επίπεδο γεών, το 30% καλύπτονται από αυτό το μέτρο. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στο ελεγκτικό συνέδριο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ως φρένο για την απερίμωση της α, υπαίθρου. Γιατί ένας γεωργός έχει μια τάση και ένας επιχειρηματίας έχει μια τάση να παράγει περισσότερο. Αυτή η εντατικοποίηση της γεωργίας είναι όμως κατά είναι κατά της γεωργίας. Στην έκθεση επίσης λέμε ότι οι άμεσες πληρωμές είναι το 30% των πληρωμών. Είναι μία στήριξη του εισοδήματος, γιατί οι γεωργοί πρέπει να κάνουν μία σειρά από πράγματα, μία σειρά από εργασίες, και το να παραιτηθούν από την υπερβολική παραγωγικότητα τους φέρνει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους ε, υπόλοιπους ε, μη ευρωπαϊκούς ε, γεωργούς. Επομένως αυτές, αυτή η βοήθεια που δίδεται είναι απαραίτητη. Γιατί ο γεωργός έτσι έχει ένα ελάχιστο εισόδημα να βασιστεί. Για να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες με τις οποίες παράγουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση ότι όλες οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να συνδέονται με το πρασίνισμα δίνει μία προστιθέμενη αξία σε σχέση με την οικοαιρεσιμότητα για να αντιμετωπίσουμε την, τον ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την ε, γεωργική πολιτική στις ε, κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ε, και στον άκρατο ανταγωνισμό που είναι κατά του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αυτός είναι ο στόχος των μέτρων αυτών. Πέρα από την ακρίβεια των αριθμητικών στοιχείων που μας δίνει το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστούμε κύριος Γερμπλόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για τις ε, παρουσιάσεις και τις ε, δύο αυτές εκθέσεις, και όχι μόνο για αυτές τις δύο, αλλά και εκείνη που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα για την κοινή γεωργική πολιτική. Και αυτή μετέφερε ένα μήνυμα καταστροφής ότι όλο το οικοδόμημα της κοινή γεωργικής πολιτικής ουσιαστικά δεν συνάδει με τους αρχικούς στόχους. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί αυτή τη φορά όντω είναι ε, έγκαιρη η ανάλυση τους. Γιατί την περασμένη φορά, όταν υπήρξε μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, σε περισσότερες εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, δημοσιεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Οπότε σας συγχαίρω γι' αυτό. Για μένα το μήνυμα είναι σαφές. Έχουμε μέτρα περιβαλλοντικής διάστασης, Έχουμε πολλούς περιβαλλοντικούς ε, στόχους που συνδέονται με, τα, με τους δημόσιους πόρους ε, που δαπανούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των στόχων και των ε, δαπανών. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Εξέτασα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις δύο εκθέσεις και ουσιαστικά δεν υπάρχουν σχόλια λένε ότι εντάξει το εξετάζουν και θα επανέλθουν με σχόλια στην τελική τους πρόταση για την επόμενη κοινή γεωργική πολιτική. Και αυτό μου θυμίζει την περασμένη φορά, όπου η Επιτροπή ουσιαστικά δεν άκουσε ε, τα δεδομένα, τα στοιχεία που τους μετέφερε το ελεγκτικό συνέδριο. Για μένα είναι απλά τα πράγματα. Έχεις ένα στόχο, βρίσκεις τα κονδύλια και τα δαπανάς για να πετύχεις τους στόχους. Όταν βλέπουμε ότι δεν πετυχαίνουμε τους στόχους με την πολιτική ή με τους πόρους που έχουμε δαπανίσει, τότε αλλάζουμε την πολιτική. Ε, αυτό το τελικό συμπέρασμα ποτέ δεν έχει βρεθεί στην Ευρώπη ξοδεύουμε δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων για το πρασίνισμα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να παροτρύνω το Ελληνικό συνέδριο ε, να είναι ακόμα πιο ξεκάθαροι στις δηλώσεις τους, να μην μας ανταλλάσσουν τα λόγια τους και το μήνυμα να φτάσει όχι μόνο στο κτίριο Μπελεμών, αλλά και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, αλλά και στις ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί μιλώντας με συναδέλφους, βλέπω μεγαλύτερη έμφαση στο, στην πεπατημένη και στα πράγματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, παρά στους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και στα στοιχεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να ρωτήσω την Πρόεδρο αν θα μπορούσαμε να λάβουμε και ένα σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν την υποβολή των νέων προτάσεων που να είναι πιο λεπτομερείς Να μπαίνουν δηλαδή συγκεκριμένα ε, στο, να σχολιάζουν τις εκθέσεις του Ελληνικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κυρία Σκαρεπίρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. από τις ε, κάτω χώρες να μεταφέρουν διαφορετικό μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με, τις, ε, με τους πολιτικούς στόχους, τους πόρους ε, και την πολιτική. Θα πρέπει η πολιτική να είναι εφαρμόσιμη. Ευχαριστώ τους ομιλητές γιατί από το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Και εγώ από την Ολλανδία προέρχομαι και βλέπω πολλού νέου γεωργού που δεν θέλουν να σταματήσουν επειδή δεν έχουν γεωργική εκμετάλλευση και δεν θέλουν να επενδύσουν στην καινοτομία και ε, στο νερό και στον, ε, στην ατμόσφαιρα. Όμω το πρόβλημα είναι ότι πάντα ε, είναι ασαφή η πολιτική. Ο Γιωργός είναι επιχειρηματίας Και εδώ στρέφομαι στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Πώς τα μετράμε όλα αυτά. Είναι τόσο περίπλοκη η διαδικασία ε, και οι γεωργοί είναι διαχειριστές ε, της υπαίθρου, έτσι γενικά, που τελικά τα στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. αν λάβετε υπόψη την πολιτική μας για το νερό, τη γη και την ατμόσφαιρα, την, ε, τις προτάσεις μας για την κλιματική αλλαγή ε, και τις μελλοντικέ μας πολιτικές ε, για το διοξείδιο του άνθρωπου και το καθεξής, τότε θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως έρθει η ώρα για ένα πραγματικό πρόγραμμα σε κάθε χώρα με τους πραγματικούς γεωργούς επιχειρηματίες. Γιατί εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τους γεωργούς, όχι να το αφήσουμε στις πολυεθνικές γιατί εκεί έχει να κάνει με τις επενδύσεις και το ποσοστό κέρδους. Ενώ εδώ βρισκόμαστε στο κέριο σημείο, γιατί τώρα βλέπουμε ότι διώχνουμε τους γεωργούς και δίνουμε στο πιάτο την ύπεθρο για τις πολυεθνικές. Και τότε θα χάσουμε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Γιατί τα στατικά είναι σωστά, όμως ε, στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριος Ντες. Ε, ευχαριστούμε για τις δύο παρουσιάσεις. Ε, να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως την κυρία Φωσκεύση. Ε, λοιπόν, θα ήθελα, επειδή έχω ήδη τοποθετηθεί στην Επιτροπή Γεωργίας, να πω ότι στα 14 χρόνια ε, που είμαι εδώ πέρα ποτέ δεν είδα ε, τόσο κακή έκθεση από πλευράς ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Ήδη και ο χρονισμός από το 2016 βλέπουμε πόσο ανεπιτυχές ήταν το screening για τα δύο χρόνια. Το 2015 ήδη τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν σε κατευθυντήριες ε; και το 2016 δυσκολεύτηκαν πάρα πολλά κράτη-μέλη για να τις εφαρμόσουν. Δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτημα για το 2016 ε, και βλέπετε λοιπόν πόσο κακά ήταν τα αποτελέσματα του screening. Διάβασα δύο φορές ε, αυτήν την έκθεση και βλέπουμε ότι απευθύνει κριτικές ε, το ελεκτικό συνέδριο για τις δαπάνες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γραφειοκρατία. Εμείς θέλαμε, ήταν πολιτική βούληση να προωθήσουμε την ε, βιοοικονομία. Ε, εμείς ε, πήραμε πολιτική απόφαση να μιλήσουμε για το πρασίνισμα. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιε παρατηρήσει μετά το ελεγκτικό συνέδριο και μας λέει ότι όλε αυτές οι διατάξει είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές και δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτέ τι απαιτήσει. μα εμείς το αποφασίσαμε. Επίσης δεν αξιολογήσαμε ε, την κατάσταση διότι παραγνωρίζουμε τη σημασία της διάβρωσης, παραδείγματος χάρη του εδάφους, που, γιατί μετά δεν είναι μια γη και μιλάμε, μιλάτε για τη μείωση ε, του εμβαδού της ε, καλλιεργήσιμης γης ε, και δεν μετράτε ούτε σπλημμύρες ούτε τη διάβρωση γης, ούτε κανένα τέτοιο παράγοντα. Υπάρχουν και άλλα σημεία που δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι ε, πρότεινε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έπρεπε εμείς να έχουμε κινηθεί. Ε, συγγνώμη, κατάρα δηλαδή, θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο όταν προτείνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε να αποφανθεί. Εμένα δεν με νοιάζει τι πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιηθεί το ελεγκτικό συνέδριο νωρίτερα γιατί εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό όργανο και έχουμε μια πολιτική βούληση αλλά τη βασιζόμαστε για τι αποφάσει μα ε, στι πληροφορίε ε, που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, πως ε, για την εφαρμογή όλα αυτά έχουν σημασία. Ε, δεν λέγαμε, θέλουμε να μειώσουμε την, το εμβαδό της καλλιεργής γης, να περιορίσουμε τις γεωργικές μετάλλευση 40 εκτάρια. Δεν γίνεται όμως σε χώρες όπως η Γερμανία. Μπόρεσα λοιπόν, έπρεπε να αποσύρουμε διάφορες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μόνο και μόνο λόγω μεγέθους. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και όταν μιλάμε για το screening, στα κράτη-μέλη και ε, όταν βλέπουμε το ότι έχει 600 ευρώ στον πρώτο πυπηλόν και μετά έρχεται το πρεσίνισμα και παίρνει 80 ευρώ ε, και παίρνει 60 ευρώ ένα εκτάριο ε, και μετά δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση ας πούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις του πρασινίσματος μέσα στις εκθέσεις. Δηλαδή ο ένας παίρνει 18 ευρώ και άλλος παίρνει 180 ευρώ και αυτά είναι άμεσα αποτελέσματα του πρασίνισματο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ε, αυτό είναι σκουπίδι για μένα. Εγώ για τίποτα άλλο δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσω αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνέδριου. Ευχαριστούμε κύριε Εντές, ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τη, Δελικό συνέδριο για την έκθεση. Θέλω να σχολιάσω διάφορα ζητήματα. ναι, για το πρασίνισμα είχαμε την γνωμοδότηση τη, της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν θα είμαι τόσο σκληρός όσο ο Άλμπερτες, αλλά ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές έκτακτες περιπτώσεις και εξαιρέσεις. Παραδείγματο χάρη στη βασική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω γιατί επέμεναν για το εμβαδό τη ε, ε, βασικής εκμετάλλευσης ε, γιατί το προσδιορίστηκε και γιατί είχαμε όλες αυτές τις εξαιρέσεις δηλαδή ισοπαίδωσαν το σύστημα μετά η αμυξισπορά για ποιο, για, για λόγο πρέπει εμείς να τα ρυθμίσουμε αυτά το κάνει ο κάθε γεωργός αυτόματα Υπάρχουν περί, ε, ένα, ένα μέρος των εκμεταλλεύσεων δεν καλλιεργείται. Όταν μιλάμε για το 15% της ε, καλλιεργήσιμης γης, ε, δεν μπορούμε ξέρω εγώ, να χρησιμοποιήσουμε τα λοιπάσματα, τα παρασιτοκτόνα. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί τα πρότεινε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο εκ των υστέρων μας εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θέμα μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί τα κράτη-μέλη πολέμησαν τόσο πολύ το πρασίνισμα που τελικά δεν έμεινε τίποτα από αυτό. Ε, μιλάτε για την απώλεια της ε, βιοπικιλότητας. Ε, βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Φαίνεται από τις μελέτες και το αντίθετο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα χημικά προϊόντα. Θέλω να ρωτήσω εγώ το ελεγκτικό συνέδριο. Εσείς Πώς βλέπετε τώρα τις προτάσεις ε, του Επιτρόπου Χόγκαν, δηλαδή να εκπονούν τα σχέδια τα ίδια τα κράτη-μέλη και να θέτουν τους στόχους και να κάνουν την αξιολόγηση, να μεταβάσουν δηλαδή περισσότερη εξουσία στα, στα κράτη-μέλη. Πώς θα τις αξιολογείτε αυτές τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όπως είναι ε, τώρα η κατάσταση δεν αποφασίζουν τίποτα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ε, σας δικαιώνω εγώ σε πάρα πολλά σημεία, αλλά όταν τα λεφτά βγαίνουν από τον δημόσιο κορβανά, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τελικά τα αποτελέσματα της δράσης μας. Ε, δεύτερον, κύριε Βοσανιώσκη, μας είπατε ότι ναι, βεβαίως είναι υπερβολικές αυτές οι διοικητικές ρυθμίσεις ε, με το που υποβάλλει. Δεν προτολμάει κανένας να υποβάλει έτοιμα γιατί λόγω γραφειοκρατίας και όντως πρέπει κάτι να κάνουμε. Όμως, ε, χειροτέρευσαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε πόσο καταστροφική είναι η κατάσταση. Στο δείξατε τα στοιχεία που μας δώσατε και έχετε το δεύτερο και το τρίτο πυλώνα και ε, όλα τα σχέδια του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ε, υπονομεύονται από την ε, καταστρεπτική γραφειοκρατία. Πολύ ωραία. Κάντε μας για καμιά συγκεκριμένη πρόταση. Πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτά. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε για τα νέα προγράμματα πώς μπορούμε να έχουμε ασφάλεια δικαίου και για την ε, διοίκηση, για τις αρχές ε, και για τον ε, τόντα, ε, πώς θα το καταφέρουμε αυτό χωρίς να ε, υπονομεύουν τα προγράμματά μας η γραφειοκρατία μας. Ε, είπατε ότι χαθήκανε 19 εκατομμύρια εκτάρια γης. γιατί, ξέρετε, να μας πείτε τι, γιατί δεν υπάρχει αυτή η καλλιεργήσιμη γη, τι τα χτίσανε, έγιναν οικόπεδα, τι έγινε. Στην τελευταία εκδοχή της κοινή γεωργικής πολιτικής προσπαθήσαμε εμείς να ενθαρρύνουμε τη γεωργία και να συμμετέχουν και οι νέοι. Ξέρετε το εισόδημα του γεωργού υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Οπότε ε, τα φορολογικά κίνητρα της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν βιώσαν την κατάσταση ε, και το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, διότι φεύγουν από την ύπεθρο οι νέοι γεωργοί γιατί δεν έχουν ε, τα απαιτούμενα ε, χρήματα για να επιβιώσουν, δεν είναι ε, το εισόδημά τους ε, επαρκές. Και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βλέπετε τι παίρνουν οι γεωργοί, βλέπουν τι, τι παίρνουν... Η γαλακτοπαραγωγή, παραδείγματο χάρη, είναι 100% αποσυνδεδεμένη από τις άμεσες πληρωμές κοινή γεωργικής πολιτικής. Λοιπόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα προστοζήνια τους γεωργούς, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάθε αξιολόγηση βασίζεται σε πολλά διαφορετικά στοιχεία και κριτήρια, τα οποία μπορεί κάποιος να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Αλλά νομίζω ότι στην ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ θα πρέπει κανείς ένα και μόνο πράγμα. Ότι η γεωργία αφορά την παραγωγή τροφίμων, αλλά και άλλα πράγματα, άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες. Η γεωργία συμβάλλει στην παραγωγή και διατήρηση των κοινών μας πόρων, για παράδειγμα το περιβάλλον. Με το πρασίνισμα θέλουμε ακριβώς ε, να υποστηρίξουμε αυτόν τον ε, κοινό πόρο. Βλέπουμε λοιπόν ορισμένες τάσεις ε, που μας ανησυχούν, κάποιοι δείκτες, όπως ο αριθμός των πτηνών, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Όμως, θα ήθελα να έχουμε κατά νου αυτόν τον πολυπαραγωγητικό ε, χαρακτήρα της γεωργίας. Γιατί η γεωργία μας δίνει δημόσια αγαθά, τα οποία θα πρέπει να κοστολογούνται επαρκώς. Εφόσον θέλουμε να συνεχίσει η Γεωργία να μας παρέχει αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε ε, οικονομικές ε, συναλλαγές υπέρ της Γεωργίας. Αυτό βέβαια ίσως να ήταν πιο εύκολο αποδεκτό από όλα τα διαφορεμένα μέρη. Να θυμάστε όμως ότι είχαμε στήριξη με βάση την τιμή και είχε δεχθεί δρυμύτατη κριτική. Τώρα η στήριξη δίνεται ανάλογα με το εισόδημα. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς για να κάνουν ορισμένες αλλαγές. Στηρίζουμε λοιπόν ε, τους γεωργούς ή πολύ απλά τους πληρώνουμε τους γεωργούς για να το πούμε με απλά λόγια για να μας ε, ε, παραδώσουν ε, δημόσια αγαθά. Είχαμε την δήλωση του 1996 και την δήλωση του 2016 που μιλούσε ακριβώς για τον ε, πολυπαραγωγικό χαρακτήρα της γεωργίας σε σχέση με τον ε, τόπο κατοικίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης η γεωργία συμβάλλει και στην ε, πολιτιστική μας κληρονομιά. Είτε αυτή είναι ηλική είτε άειλη. Νομίζω ότι όλες αυτές οι πτυχές λοιπόν θα πρέπει ε, να επισημανθούν. Και από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτή τη διάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, λειτουργίες και κατά πόσο τιμολογούνται σωστά, κοστολογούνται σωστά, νομίζω πως όχι, δεν πληρώνουμε αρκετά για αυτές τις λειτουργίες, όπως προκύπτει και από την, ε, τις επιστημονικές μελέτες. δεν δίνουμε μεγάλα κίνητρα, οικονομικά κίνητρα στη Γεωργία. Ε, κάπως αντισταθμίζουμε συγκεκριμένες δαπάνες των Γεωργών ε, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Και κάτι τελευταίο. Δεν ε, συμβαίνει αυτό μόνο με την ευρωπαϊκή γεωργία, ότι δέχεται δηλαδή οικονομικά κίνητρα ε, με αντάλλαγμα συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Για παράδειγμα, και στη Βραζιλία υπάρχει ανεπτυγμένη γεωργία και εκεί λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αν θέλουμε να, να διατηρήσουμε τη γεωργία μας, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία. Από τη μία πρέπει να δώσουμε αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς και από την άλλη θα πρέπει να συνεχίσουν οι γεωργοί να παρέχουν αυτά τα δημόσια αγαθά που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο τέλος του καταλόγου. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ιδάλλως, να δώσω το λόγο στους συζητητέ. Ο κύριος Γέρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα σας τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω με τα ερωτήματα του κ. Γερμπράντη. Είπε ότι βρήκαμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ στόχων και δαπανηθέντων πόρων. Αυτό ισχύει σε ένα βαθμό, όμως το πραγματικό μας έβριμα είναι ότι δεν υπάρχουν στόχοι. Εφόσον δεν υπάρχουν στόχοι, δεν να... Δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, δεν μπορούν να υπάρξουν δείκτες ε, και να δούμε πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα μέτρα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο λογιστικό έλεγχο. Δεν ξέρουμε πώς, ποια θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση προς ε, την βιοπικιλότητα, προς ε, τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου και το Για μας αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν έχουμε αφετηρία. Ποιος ήταν ο στόχος μιας πολιτικής. Μετά πώς μπορούμε να κρίνουμε το αποτέλεσμα και αν διοχετεύτηκαν σωστά οι πόροι. Συζητήσαμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως τι θα πρέπει να βελτιώσουμε, τι εννοούμε με τη βελτίωση της κλιματικής απόδοσης για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να βελτιώσουμε τους δείκτες μας ή απλώς ε, να περιορίσουμε την πτώση ή να σταματήσουμε την πτώση του περιβαλλοντικού δείκτη. Αλλά αυτό δεν είναι σαφές. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα του ελέγχου. Η κυρία Γιούσο τώρα. Ό,τι είπατε ισχύει. το νόημα δηλαδή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Όμως μετά έχουμε τους στόχους και από τους στόχους πάμε στα μέτρα. Τα EFAs λοιπόν, πολλές φορές ε, το θίξατε αρκετοί. Είπαμε στην, στην έκθεσή μας ότι οι γεωργοί ήδη έχουν δώσει το διπλάσιο ε, αριθμό EFA σε σχέση με το greening. Δεν είναι δηλαδή το πρασίνισμα που δημιουργεί την οικολογική, την περιβαλλοντική απόδοση. Οι γεωργοί τα πήγαιναν πολύ καλύτερα και πριν από την υλοποίηση αυτού του μέτρου. Όταν λοιπόν πρέπει να δούμε τι ακριβώς πετυχαίνουμε με το πρασίνισμα, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα υπάρξει μία αλλαγή. Η αλλαγή θα προκύψει εξαιτία του πρασινίσματος ή εξαιτία κάποιε άλλη προαιρετική δράση που αναλαμβάνουν οι γεωργοί. Ότι βελτιώνουν την τεχνογνωσία του ή ακόμα και την αντίληψη που έχουν για τι περιβαλλοντικέ απαιτήσει από αυτέ που του ε, επιβάλλει το πρασίνισμα. Ο κύριος Δές έθεσε μία σειρά ερωτήματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα ερωτήματα που μας ε, στείλατε. Ήδη έχουμε προετοιμάσει τις απαντήσεις και θα τις στείλουμε σύντομα και πιστεύω ότι έτσι θα διευκρινιστούν πολλές ε, παρανοήσεις ε, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της εκθεσής μας γιατί έχουμε ακολουθήσει όλα τα διεθνή ε, πρότυπα λογιστικού ελέγχου. Εξετάζουμε το τι ακριβώς στόχο θέλουμε να πετύχουμε με το πρασίνισμα, όχι το τι κάνουν οι γεωργοί, σωστά ή λάθος. Για να απαντήσω εν συντομία κάποιες από τι ερωτήσει, σας και μετά λεπτομέρειε θα τα λάβατε γραπτός είπα ότι για τα EFAs οι γεωργοί τα πηγαίνουν καλά, έχουν διπλάσια έφαση σε σχέση με την ε, προϋπόθεση. ακόμα και για το πρασίνισμα. Λέμε ότι στην Πολωνία ήδη το 30%, οι γεωργοί έχουν 30% παραπάνω έφαση από ό,τι απαιτείται από το πρασίνισμα. Ακόμα και αν μιλούμε για το έτος 2016, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε το συμπέρασμα ότι η πολιτική έχει πετύχει τον α ή τον β στόχο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι ε, είναι μάλλον απίθανο να βελτιώσει σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση. Ξέρετε όμως πολύ καλά, είπε και ο κύριος Ράινσταν. Θα ήταν ε, ανόητο να, περι... να περιμένει κανείς ε, διαφορετικά αποτελέσματα εάν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες δράσεις. Εάν δεν αλλάξουμε λοιπόν τίποτα, παρόλο το βρασίνισμα, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Για τα catch crops, εμείς ε, εστιαστήκαμε ε, στην περίοδο πριν από, τις, ε, από τον κανονισμό, όμως και πάλι αυτές οι καλλιέργειες αφορούσαν μια περίοδο 8 εβδομάδων μόνο, όχι για όλο το χειμώνα. Για τις ενδιάμεσες καλλιέργειες. Εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονε, αλλά αντλήσαμε στοιχεία από άλλες μελέτες εμπειρογνωμόνων. Θα τα δείτε στη δική μας έκθεση και θα απαντήσουμε, στι απαντήσει μα μάλλον θα βρείτε και αυτό. Ποιε μελέτες χρησιμοποιήσαμε. Αν δείτε και τον δεύτερο ε, πίνακα, και οι Ολλανδοί επιστήμονες είχαν πει να μην βάλουμε τις ενδιάμεσες καλλιέργειες εκεί, όπως ε, είχε προταθεί με το πρασίνισμα. Μετά ο κύριος Χάουσλινγκ με ρώτησε γιατί να μην δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Εναπόκειται στους πολιτικούς να αποφασίσουν ποιος θα φέρει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνη. Εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα αυτή η προσέγγιση, όμως τονίζουμε, και αυτή είναι και η σύσταση προς τα κράτη-μέλη, ότι θα πρέπει να δείξουν ότι τα ε, μέτρα που θα επιλέξουν θα έχουν όντω τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα συμβάλλουν γενικά στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου. Γι' αυτό, ακόμα και αν η Επιτροπή έλεγε, εντάξει, τα κράτη-μέλη θα έχουν περισσότερε αρμοδιότητε να επιλέξουν ορισμένα μέτρα ή ε, κατηγορίε EFAs, περιοχών οικολογική εστίαση, και πάλι όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ελέγχει και να υιοθετεί τα εθνικά προγράμματα που θα πάρουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που επιλέγονται όντω ε, βελτιώνουν το αποτέλεσμα. Ένα άλλο ερώτημα, ή έγινε μια συζήτηση του κ. Γκριπς, λέει ο Μίλτης, και είπατε ότι τα δημόσια αγαθά, η παροχή δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να χρηματοδοτείται. Σωστό όμως. Το βασικό ερώτημα είναι πόσα λεφτά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ποιο θα παίρνει αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν είναι θέμα που θα το απαντήσει ένα λογιστή. Όταν διαμορφώνετε τη λογική παρέμβαση θα πρέπει να ξεκινήσετε από τους στόχους, ε, να καθορίσετε τους δείκτε, ε, να επιλέξετε τα μέτρα και να αποφασίσετε ε, πόσα λεφτά δαπανώνται. Και εμεί, μετά, ως ελεγκτές, ως λογιστές, ελέγχουμε το κατά πόσο τα λεφτά τα οποία δαπανώνται δαπανώνται για τον στόχο ΑΒΓ, ας πούμε, και κατά πόσον υλοποιείται. Ε, πάντως, όταν διαμορφώνεται τη λογική της ΚΑΠ, εκεί θα πρέπει να δούμε ποιος ε, παίρνει τα λεφτά για να παράγει όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και για να έχει κάποιες περιβαλλοντικές επιδόσεις η ΚΑΠ. Να κάνει κάποια πράγματα υπέρ του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά, τη μητρική μου γλώσσα. Ε, Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις, λέει ο κύριος Βολτσόφσκι, και για τα σχόλια. Με μεγάλη χαρά βλέπω την κατεύθυνση την οποία, και την τροπή την οποία πήρε η συζήτηση. Δείχνει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ο κ. Ξύπ, ο κ. Μπλάντινγκ μίλησαν για την πολυλειτουργική φύση της γεωργίας. Δεύτερον, αυτά που είπα και εγώ και ο συνάδελφος σήμερα, ήθελα να σας επιστήσουν την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο διαπιστώνουμε. Εάν το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι η απλή συνέχεια της ε, σημερινής κατάστασης, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να συμφιλιώσουμε την ΚΑΠ με την περιβαλλοντική πολιτική. Εάν οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι μικροί γεωργοί, οι μικροί καλλιεργητές εξαφανίζονται και αν βλέπουμε όλο και περισσότερο μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιούμε τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους. Θέλουμε να το εντοπίσουμε αυτό το θέμα, να το υπογραμμίσουμε. Βεβαίω οι πολιτικοί πρέπει να αποφασίσουν πόσε ε, γεωργικές εκμεταλλεύσει θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2030, Φερρυπίν. Όχι του χρόνου, όχι αύριο μεθαύριο, το 2030. Το σκεφτόμαστε αυτό το θέμα. Έχουμε μια μακροπρόθεσμη κλιματική πολιτική και είναι πολύ θετικό βεβαίως το να καθορίζουμε τους στόχους μας μακροπρόθεσμα αλλά τη γεωργία δεν τη βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Δεν έχουμε αυτό το όραμα. Δεν ξέρουμε πόσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, το 2050. Μέσα σε 10 χρόνια χάσαμε 4 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πόσες θέλετε να έχουμε, 5 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ή λιγότερες. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο το οποίο να μιλάει για αυτά τα πράγματα και θα ήταν απαραίτητο κάτι τέτοιο. Όσο μεγαλύτερε εκμεταλλεύσει, είναι πολύ πιο δύσκολο να παντρέψουμε αυτέ τι λειτουργίε μια μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση με τι περιβαλλοντικέ ανάγκε. Το γεγονό ότι εξαφανίζονται οι μικρέ εκμεταλλεύσει, ότι ο γεωργικό πληθυσμό γυράσκει, ότι οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί δεν έχουν κάποιον να του διαδεχθεί, δεν έχουν παιδιά που να θέλουν να κάνουν το ίδιο επάγγελμα. Αυτό είναι ένα μονόδρομο. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να βλέπουμε μια πιο έτσι, δυναμική γεωργία, αλλά μην ξεχνάμε και το περιβάλλον. Και χαίρομαι που το εντοπίσατε στις παρεμβάσεις σας. Δύο ευρωβουλευτές μίλησαν επίσης για την ε, δική τους ε, πραγματικότητα στη δική τους ε, χώρα. Σε ποιο βαθμό θέλουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και σε ποιο βαθμό θέλουμε μια εθνική γεωργική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση πραγματικά ποικίλει. Στην Τσεχία, ας πούμε, το μεσαίο μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 130 εκτάρια. Ενώ στην Πολωνία, ας πούμε, είναι λιγότερο από 10 εκτάρια. Επίσης, έχουμε πολύ διαφορετικές καταστάσεις ότι αφορά την ηλικία του γεωργικού πληθυσμού. Στην Πορτογαλία, ας πούμε, το 50% των γεωργών είναι 65 και πάνω χρονών. Έχουν φτάσει δηλαδή στο συνταξιδοτικό του όριο. Σε πολλές χώρες η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη βεβαίως. Στην Πολωνία, Φερρυπίν, ή στην Αυστρία, στη Γερμανία. Η ηλικία του γεωργικού πληθυσμού είναι τελείως διαφορετική. Είναι πολύ πιο νέοι η γεωργοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως προτείνει τα ίδια πράγματα, τις ίδιες δραστηριότητες και τα ίδια κίνητρα σε όλους τους γεωργούς και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε το ίδιο φάρμακο και την ίδια συνταγή, ας πούμε, ε, για όλες τις αρρώστιες, για όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Θέλουμε μια πιο ευέλικτη γεωργική πολιτική. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό θέμα που πρέπει να συζητήσετε και να αποφασίσετε. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ο κύριος Χόισλινγκ ε, έθεσε ένα τέτοιο ερώτημα. Μιλάμε για 19 εκατομμύρια εκτάρια. Είναι μια τεράστια έκταση. Είναι περίπου το μισό της έκτασης της Γερμανίας. Και δεν ξέρουμε μέσα σε μια δεκαετία που εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε τι συνέβη, πώς φτάσαμε εκεί. Έχουμε κάποια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι αυτή είναι η μείωση της γεωργικής γης με βάση τα στοιχεία, τα δηλωμένα στα πλαίσια της ΚΑΠ. Θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με αυτή τη γη. Δεν ε, εξαφανίστηκε στο υπερπέραν, αλλά δεν δηλώνεται πια ως γεωργική γη, ως γεωργική έκταση όλη αυτή η έκταση. Επίσης, να σας πω ότι θα ετοιμάσουμε ακόμα ένα έγγραφο, μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και θα το ετοιμάσουμε αφού δούμε την ειδική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ελεκτικό Συνέδριο έχει συντάξει πάρα πολλές νομοδοτήσεις ήδη και νομίζω ότι ο κ. Γκερμπράντι είπε ότι είμαστε καλύτερα εφοδιασμένοι και προετοιμασμένοι για να συζητήσουμε το μέλλον της ε, ΚΑΠ. Σαφώς είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι σε σχέση με την περασμένη φορά. Εγώ στο, το, την προηγούμενη φορά ήμουν ευρωβουλευτής και θυμάμαι ότι δεν είχαμε πολλές πληροφορίες. Δεν είχαμε τόσες όσες έχουμε σήμερα. Επίσης, Θα ήθελα επ' ευκαιρία να σας μιλήσω λιγάκι για τις μελλοντικέ δημοσιεύσεις